el señor presidente. Buenas tardes, colega. Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. άρχε τη συνεδρία έχουν διανεμηθεί τα συνοπτικά πρακτικά της εσύνης συνεδρίας. Δεν έχει κανείς κανένα σχόλιο να κάνει στα πρακτικά. Θεωρούνται και